La séance est ouverte. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Φαντάζομαι δεν έχετε παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη και μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ανακοινώσεις του Προέδρου δεν υπάρχουν. Οπότε ερχόμαστε στο ένα και μοναδικό θέμα της συνεδρίασής μας που είναι η παρουσίαση του εγγράφου προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα έγγραφο προβληματισμού που θα μας παρουσιάσει ο Επίτροπος Έτιγκερ, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους. Φαντάζομαι θα μιλήσετε και για τη συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση Μόντι για τους ιδίους πόρους. Σας ευχαριστούμε θερμότατα κύριε Επίτροπε που εκφράσατε την επιθυμία ε, να έρθετε εδώ για να μας παρουσιάσετε αυτό το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έρχομαι χαρά εδώ το έγγραφο αυτό προβληματισμού είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ένα αρκτήριο λάκτισμα που θέλουμε να δώσουμε, η βάση που θέλουμε να ορίσουμε για μια επικοδομητική σειρά συναδελφικών ανταλλαγών απόψεων για την πολιτική του προϋπολογισμού, τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσεχή δεκαετία. Σήμερα συστήθηκε και εγκρίθηκε το έγγραφο αυτό στην Επιτροπή, στη συλλογική της μορφή, με την κυρία Κρέτσου αρμόδια για την ε, πολιτική συνοχή. Και θα ήθελα να σας αναφέρω το κύριο περιεχόμενο και τη στρατηγική εν συντομία και βέβαια θα επεκταθώ και περιμένω και τις ε, απόψεις, της προτάσεις σας, τις επικρίσεις σας. Έχουμε δύο ή τρία κενά επί της ουσίας, τα οποία είναι ουσιαστικά ουσιώδους σημασίας για την επόμενη δεκαετία. Ανεξαρτήτως της περίοδου που θα κρατήσει αυτό, ξέρουμε ότι από εδώ και μπρος δεν θα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Βρετανοί και δεν θα συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Έχουν το 16% των εσόδων οι Βρετανοί και παρά την σοβαρή επιστροφή που έχουν, έχουν χαρακτήρα καθαρού χορηγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 10-11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπουμε την μεγάλη ευθύνη αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία που μας προσφέρεται με τη νέα καθήκοντα αλλά και τα νέα προβλήματα τα ευρωπαϊκά να τα λύσουμε με ευρωπαϊκό τρόπο. Είναι απαραίτητη λοιπόν η δημοσιονομική πόρη για την ικανοποίηση αυτών των καθηκόντων στα θέματα του προσφυγικού, της μετανάστασης, των προστα... της προστασίας των συνόρων, του ελέγχου των συνόρων, της τρομοκρατίας. του σημαντικού τομέα της εξωτερικής ασφάλειας, της άμυνας, αλλά και της εσωτερικής ασφάλειας. Μπορεί βέβαια κανείς να συζητήσει το ύψος των πόρων που θα χρειαστούν για να εξασφαλιστούν αυτοί, αυτά τα καθήκοντα, για να λοιπηθούν τα καθήκοντα αυτά. Αλλά πάντως διαρθρωτικά και για κάθε χρόνο θα μιλούμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτον. Ένα άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να επισέλθουμε και να καλύψουμε έχει να κάνει με, την, ε, με τους εξωτερικούς πόρους το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτυξιακής Βοήθειας να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και εδώ οι προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύονται όπως ενισχύεται και η σαφήνεια του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Δύο-τρία λοιπόν αρκές με 20 δισεκατομμύρια ή και περισσότερα ευρώ το χρόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δι' η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλο μέρος του καθήκοντος να επιτελέσει, διότι εμείς θα πρέπει να επαληθεύσουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε για να καλύψουμε τα υφιστάμενα κενά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ζητήσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα έσω πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Εξυγχρονισμός, απλούστευση, απλοποίηση των προγραμμάτων μας, περισσότερη ακόμη ευελιξία μεταξύ των δημοσιονομικών ετών, των κεφαλαίων και των προγραμμάτων, των τίτλων του προπολογισμού και των ε, προγραμμάτων, ενδεχομένως μετακινήσεις πόρων, ενδεχομένως δε και σοβαρές αλλά πάντως θεμητές περικοπές. Με το spending review, την αναθεώρηση των δαπανών, έχουμε μία βάση. Και έτσι σε, ε, αυτό το κάνουμε για όλα τα μεγάλα μας προγράμματα, στον τομέα της γεωργίας, στους δύο πυλώνες, στα διαρθρωτικά ταμεία, ταμεία συνοχής, κοινωνικό ταμείο, στο μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη, στον ορίζοντα 2020, όπως και στο ΕΤΣΕ, το σχέδιο Juncker. Άπαξ και ολοκληρωθεί αυτή η επισκόπηση και σε αυτό ζητούμε τη δική σας συμβολή, και πραγματογνωμοσύνη της Επιτροπής των Προπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, με τους βουλευτές οι οποίοι γνωρίζουν στην κάθε περιφέρεια πώς λειτουργούν και τι αποτελέσματα φέρνουν τα προγράμματα, αλλά έχουν εντοπίσει και τις ανάγκες για επενδύσεις. Η δική σας λοιπόν συμβολή είναι πολύ σημαντική και εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να ε, ενισχυθεί η δράση του Ευρωπαϊκού προπολογισμού, η καλύτερη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπή, η πιο αποτελεσματική εκτέλεση και πρέπει να αναλάβουμε και εμεί μέτρα για να είμαστε και αξιόπιστοι και να μπορούμε, απευθυνόμενοι στα κράτη-μέλη, να μιλήσουμε για μια γνήσια μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών δομών. με τα τρία αυτά κενά που μας ε, περιμένουν με το Brexit, επί παραδείγματι, διότι ο καθαρός χορηγός ε, στον προπολογισμό, στον δεν θα είναι διατεθειμένος να αφήσει να χαθούν πόροι και να υπολείπεται ο προπολογισμό λόγω της αποχώρησης της Βρετανίας, άρα θα χρειαστούν και περισσότερα χρήματα από τους 27 που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και περικοπές. Επομένως, μια αναδιανομή μεταξύ περισσότερων πόρων αφενός, αλλά και περικοπών, σε αναλογία 50 προς 50, 60 προς 40, 40 προς 60. Στα νέα καθήκοντα τώρα που αναλαμβάνουμε, όπως είναι η άμυνα, έχετε λάβει το έγγραφο προβληματισμού για την άμυνα με ένα δισεκατομμύριο για κάθε χρόνο στο προσχέδιο δημοσιονομικό πλαίσιο και 500 εκατομμύρια στην έρευνα στον χώρο της άμυνας. Και αν αναλαμβάνουμε νέα καθήκοντα για να απαλλάξουμε από ένα μέρος του βάρους που έχουν τα κράτη-μέλη, εξωτερικό έλεγχο που θα αναλαμβάνουμε πλέον ε, εμείς, αλλά και ταυτόχρονα θα μειώνονται οι ανάγκες για εσωτερικούς ελέγχου στα ιστορικά σύνορα, τότε αυτά τα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε εμείς αποβαίνουν προς όφελος και των κρατών μελών. Και γι' αυτό θα χρειαστούν και χρήματα. Ένα ποσό πρέπει να καλυφθεί, ένα 80% πρέπει να καλυφθεί και βέβαια ένα μικρότερο ποσοστό θα καλυφθεί από την ευελιξία και από μετατοπίσεις κονδυλίων. Το τρίτο λοιπόν κενό, η εισαγωγή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξωτερικών πόρων, ταμείων, θα πραγματοποιηθεί μόνο όμως όταν διατίθεται τα κονδύλια. Εάν ένα ταμείο δεν έχει ακόμη, δεν έχει αρκετούς πόρους, αλλά μόνο μας επιβαρύνουν περισσότερα καθήκοντα και δεν προέρχονται οι πόροι από τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν πόροι δηλαδή, αντί να έχουμε μια ισορροπία δημοσιονομική, θα οδηγηθούμε σε αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Άρα αυτό θα σημαίνει επιπλέον εισφορά πόρων από τα κράτη-μέλη για τον προϋπολογισμό, με αντίστοιχες βέβαια εξουσίες και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθήκον μου θεωρώ στο μέγιστο δυνατό να εξασφαλίσω και να αποδείξω την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και με βάση την αρχή της επικουρικότητας και θα ζητήσουμε βεβαίω και πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και την έγκριση των κρατών μελών. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καθώς στο έγγραφο προβληματισμό αναπτύσσουμε και το συλλογισμό του τι μπορεί να σημαίνει αυτή η προστιθεμένη αξία. Μπορούμε σε δημοσιονομικούς όρους να την ορίσουμε. Στο χώρο της, α, ε, της έρευνας. Εάν έχουμε να ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, ένα joint undertaking, ένα σημαντικό κοινό πρόγραμμα το οποίο δεν θα μπορεί κανένα κράτος μέλος μόνο του να ορίσει ή να επιβαρύνει μόνο μία συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο ή δραστηριότητα, τότε θα έχουμε ευρωπαϊκά, ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό, κράτη και βιομηχανία σε μια ευρεία συνεργασία, δημόσιο ιδιωτικού τομέα, τότε θα τα καταφέρουμε στην διασύνδεση μέσω του Δούναβη της Αυστρίας προς τη θάλασσα. Εάν μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συγχρηματοδοτήσουμε. Εάν έχουμε το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη ε, που θα καλύπτει 6-7 κράτη μαζί με τη Σερβία, τότε θα είναι πολύ πιο σαφής η απόδειξη της, υπεραξι... της ευρωπαϊκής αυτής προσθέμενης αξίας και πολύ πιο ε, εύκολο να αποδειχθεί. Η βοήθεια της Σερβίας μπορεί να σημάνει ταυτόχρονα και προσθέμενη αξία για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξασφαλίσει την ειρήνη ύστερα από ένα φρικτό εμφύλιο πόλεμο στα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής. Έχουμε πείσει την Σερβία να αποδεχθεί τις αξίες μας την ιστορική μας ένωμη τάξη να μην λύνει τα προβλήματα με, το, με τη δύναμη της βίας, με τα, να μην επιβάλλει θρησκευτικέ επιλογές ε, ή να κάνει θρησκευτικέ εκαθαρίσεις με τα, η δύναμη των όπλων. Και αυτό είναι με αντίκρισμα την προενταξιακή βοήθεια. Η προσθέμενη αξία του να έχουμε την ειρήνη να μην υπάρχουν πρόσφυγες, να μην υπάρχει πόλεμος, να μην υπάρχουν στρατιώτες στα κράτη αυτά, σε απόσταση δύο ώρων πτήσης από εδώ, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι σαφής η προσθεμένη αξία, έστω και αν δεν είναι μετρήσιμη σε ακριβείς οικονομικούς όρους. Και ένα ακόμη σημείο. Επαρχία, ε, χώρος της υπαίθρου, συγγνώμη, στην ε, Βουλγαρία. Υποστηρίζουμε την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής για τη μεταφορά αγαθών, για τη μεταφορά εργαζομένων και αυτό αποτελεί προσθεμένη αξία για την Ευρώπη ολόκληρη, όχι μόνο για τη Βουλγαρία. Και έτσι θεωρώ ότι εάν υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν ΑΕΠ της τάξης των 10.000 ευρώ κατά κεφαλή, έναντι εκείνων που έχουν 50.000 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και αυτό μπορεί να σημάνει ότι μικραίνουν αποστάσεις στην Ευρώπη, τότε νομίζω ότι έχουμε μια προσθεμένη αξία. Αν σταθεροποιήσουμε την εσωτερική αγορά, αν ενισχύσουμε την αγορά εργασία, βελτιώσουμε τη θέση και τι ικανότητε του εργατικού δυναμικού, εάν μειώσουμε τι πιθανότητε τη ύφεση, τότε νομίζω ότι έχουμε εξασφαλίσει προσθέμενη αξία για τους, προσ... για τους ε, πολίτες της Ευρώπης ολόκληρες και έξω από την ε, Βουλγαρία, για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και έξω από τη Σόφια. Γι' αυτό λοιπόν με συγκεκριμένα παραδείγματα θέλουμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει προσθέμενη αξία. Και αυτό μπορούμε να το συστήσουμε από κοινού. Θέλουμε με το έγγραφό μας να διατυπώσουμε την πρόταση ότι καταργούνται όλες οι επιστροφές, διότι καλό θα είναι εάν σταματήσει αυτή η επιστροφή για το Ηνωμένο Βασίλειο να μην ε, ξεκινήσουν ή να μην υπάρχουν ακόμη τέτοιου είδου επιστροφές για τους άλλου. Όλοι συμμετέχουν, όλοι επωφελούνται. Ήδη οι πόροι. Και περιμένω εδώ με πολύ ενδιαφέρον ε, τη δική σας έκθεση. Οι προτάσεις του Μάριο Μόντι θέλουμε μέσα από το έγγραφο προβληματισμού να τεθούν προς και πιστεύουμε ότι ακριβώς εκεί όπου η νομοθεσία για τα έσοδα είναι ευρωπαϊκή, όπως σε παραδείγμα στο σύστημα των ανταλλαγών εκπομπών EDS ε, για το διδοξίδιο του άνθρακα, εκεί όπου αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία ε, από τις κλιματικές αλλαγές, Κοπερχάγη, Παρίσι, Μαρακές, ευρωπαϊκή δηλαδή επιλογή ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στόχος για περιορισμό των εκπομπών για το 2030 και το 2050, ε, καθήκοντα αντίστοιχα για τη βιομηχανία μας, δικαιώματα εκπομπών που κατανέμονται και προχωρούν ε, μειούμενα κάθε χρόνο, φέρνουν έσοδα και εφόσον η νομοθεσία ανήκει σε εσά στο Κοινοβούλιο, τότε θα υπάρχουν αυτές οι ε, αυτοί οι πόροι θα πρέπει να είναι στον ευρωπαϊκό προβλησμό και αυτό είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Και πρέπει επίσης απερίφραστα να πούμε ότι το το επίπεδο που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τηρηθεί. Πρέπει να είμαστε έντιμοι όταν φύγει ένα μεγάλο και ισχυρό κράτο όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, καθαρό χορηγό, χάνονται αυτοί οι πόροι και έρχονται νέα καθήκοντα, τότε 27 κυβερνήσει τα 27 εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να είναι και διατεθειμένα να μας δώσουν περισσότερα χρήματα. Και στον κύριο Γκάιερ, ο οποίος έδωσε και τη σχετική ενημέρωση σήμερα, απαντώ ότι ναι, πρέπει τα κράτη να είναι διατεθειμένα να διαθέσουν περισσότερους πόρους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί διαθροτικά είναι υποχρηματοδοτούμενος για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει βεβαίως να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που μας οδηγούν σε ε, έλλειμμα, ούτε και πρέπει να το πράξουμε αυτό. Γι' αυτό πρέπει αντίστοιχα να αυξήσουν τις συνεισφορές του τα κράτη-μέλη και να δεχθούν μία-δύο νέες πηγές ιδίων πόρων. Σε αυτό θα πρέπει να τα πείσουμε τα κράτη-μέλη. μακρόν, επίσης συστήσαμε τον όρο της, ε, το ζήτημα της αιρεσιμότητας και όχι μόνο για τα ταμεία συνοχής αλλά για κάθε επενδυτικό πρόγραμμα. Πρέπει όταν ε, πρόκειται να εκταμιευθούν ευρωπαϊκοί πόροι να ορίζουμε κάποιους συγκεκριμένου όρους, προϋποθέσεις, όχι τεχνικές προϋποθέσεις, αλλά και οικονομικές και άλλες. Και σε αυτό μας απασχολεί η δυνατότητα να ενισχύσουμε τις περιφέρειες, να τις καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές στη δράση τους, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, την αγορά εργασίας. Και αυτό καταγράφεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στις ε, συστάσεις αναχώρα καταγράφεται αυτό άλλωστε. Και θέλουμε να βελτιωθούν οι συστάσεις αναχώρα και να αναπτύσσονται σε πιο πρώιμο στάδιο μαζί με τα κράτη και τις περιφέρειες προκειμένου να είναι δυνατή η άγκληση πόρων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Πιστεύουμε ότι το έγγραφο προβληματισμού πρέπει καταρχάς να λάβει απαντήσει από τα κράτη-μέλη τα ίδια. Και εσείς και εμείς θα αγωνιστούμε για τους απαραίτητους πόρους και τα έσοδα. Αλλά πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν και να πούν τι αξία έχει γι' αυτά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι με δεδομένες τις πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία, με τη σταθεροποίηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου, με την πρόκληση, με τις προκλήσεις που έχουμε έξω από τα σύνορά μας, μπορούμε νομίζω να προσφέρουμε επαρκή ε, επιχειρήματα προς τα κράτη-μέλη για περισσότερη Ευρώπη, για, περισ... για υλοποίηση περισσότερων καθηκόντων από την Ευρώπη και για περισσότερα έσοδα για την Ευρώπη. Εγώ στους προσεχείς εννέα μήνες θα επισκεφθώ κάθε πρωτεύουσα για να προβάλλω αυτές τις επιλογές στις κυβερνήσεις και παρακαλώ και εσάς όπου έχετε τη δυνατότητα στις περιφέρειες όπου εκλέγεστε να ασκήσετε το καθήκον σας προβάλλοντας και το κύρος σας ταυτόχρονα για να πείσετε. Και επίσης για την επόμενη δεκαετία τα δημοσιονομικά έτη του, προ... του τωρινού δημοσ... Ε, πολιτού δημοσιονομικού σχεδίου με 150 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι είτε πάντα 50 δισεκατομμύρια, χωρίς περαιτέρω δηλαδή, είτε 140 είτε 160 δισεκατομμύρια. Εδώ έρχεται η πολιτική διάστηση. Από 125 έως 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, περισσότερη Ευρώπη, περισσότερα καθήκοντα, πάμε στα 160. Λιγότερη Ευρώπη 1% ανώτατο επίπεδο 120-125 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η ψαλίδα και αυτή είναι η διάσταση στην οποία κινούμαστε. Για το χρονοδιάγραμμα. Στριφόμαστε προς την επιλογή των αποτελεσμάτων. 5 χρόνια συν 5, 5 χρόνια μόνο ή 7 χρόνια. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη θέλουν 5 χρόνια. Πολλά ε, κράτη συνοχή επιμένουν για τα 7 χρόνια στην διάρκεια του πολιτισμού του Σχεδιασμού. Εάν μπορέσουμε ε, με ευφύ τρόπο να σχεδιάσουμε τα οικονομικά μα, τα δημοσιονομικά μα για το μέλλον, μπορούμε να μιλήσουμε για 5 συν 5 χρόνια, δηλαδή 5 χρόνια σχεδιασμό με ενδιάμεση αναθεώρηση και ακόμη 5 χρόνια με τη δυνατότητα της αναπροσαρμογής και αυτό θα το δούμε μέχρι το φθινόπωρο τι θα σημαίνει το 5 συν 5. Τα 5 τα έχουμε. Το συν 5 τι σημαίνει ακριβώς. Αυτό θα είναι η, ε, το μεγάλο καθήκον να δώσουμε απαντήσεις άξιες του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και επίσης, ξέρω ότι μπορεί και δίκαια να ανυπομονείτε και θέλετε να ξεκινήσει η συζήτηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου αλλά αφήστε μας παρακαλώ να δούμε με ψυχραιμία την πραγματικότητα και τις συνθήκες. Η διαδικασία της Λευκής Βίβλου είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έγγραφα προβληματισμού τις συγκεκριμονοποιούν. Και σας παρακαλώ στο παρόν έγγραφο προβληματισμού, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, να συμμετάσχετε εντατικά στα επόμενα δύο μισή χρόνια θα είμαι στη διάθεσή σας σε κάθε επιτροπή, σε κάθε πολιτική ομάδα, σε κάθε βουλευτή χωριστά για να ακούσω το όσο το δυνατόν πιο νωρί και όσο, πιο πολύ, ε, όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά τις προτάσεις και τις θέσεις σας για να τις μεταφέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν τώρα προχωρήσει αυτή η ιστορία μέχρι τις αρχές του 2018, δηλαδή αν χρειαστεί να περιμένουμε πρώτα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, γνωρίζοντας ότι το Brexit έχει και αυτό τις καθυστερήσεις του. Στο θέμα των πόρων δεν μπορώ να πω ότι περιμένω εκκρεμότητες δημοσιονομικές στο τέλος του χρόνου, αλλά ως προς το δημοσιονομικό προγραμματισμό, το τι σημαίνει δηλαδή συγκεκριμένα το 2020, τι, θα έχουμε το 2021, τι θα μας λείπει ως πόροι σε μόνιμη βάση, τι συνέπειες θα φέρει η αποχώρηση των Βρετανών, θέλουμε να συνεχίσουμε την αναπτύξη βοήθεια στην Αφρική επί παραδείγματι ή όχι. Όλα αυτά τα ερωτηματικά πρέπει να λάβουν απόφαση. Και πρέπει να ακούσουμε τον κύριο τι έχει να πει γι' αυτά για να προχωρήσουμε μετά στο πολιτές δημοσιονομικό σχέδιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο σωστός τρόπος να εργαστούμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι το αργότερο μέχρι την άνοιξη του 2018, οπωσδήποτε πριν τι θερινέ δεκοπέ του 2018, εάν έχετε και εσεί τη διάθεση, θα είστε ενήμεροι για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Αλλά για να μην καταλήξει σε ένα αρχείο αυτή η πρόταση πρέπει να εργαστούμε όλοι πολύ εντατικά. Και ένα τελευταίο σημείο. Περιμένουμε μια εντολή από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το χρονικό παράθυρο μέσα στο οποίο εντάσσουμε αυτές τις ε, συνομιλίες. Δύο χρονικά παράθυρα έχουμε ουσιαστικά να επιλέξουμε, δηλαδή μετά τις Ευρωπα... ευρωεκλογές του 2019, δηλαδή μετά το καλοκαίρι του 2019 και την εκείνη των εργασιών της Επιτροπής σας που θα είναι το Νοέμβριο του 2019. Επομένως εκεί έχουμε από τα τέλη του 2019 έως τα τέλη του 2020 ένα χρόνο περιθώριο. Ένα χρονικό περιθώριο ενός έτους ολόκληρου. Ιδάλλως από τα τέλη του 2018 μέχρι τις ευρωεκλογέ του 2019, πάλι έχουμε ένα χρόνο στη διάθεσή μας. Και στις δύο περιπτώσεις και τα δύο χρονικά παράθυρα έχουν την ίδια διάρκεια. Η χρονική πίεση με το 2020, τα τέλη του 2020 είναι δεδομένη. Αλλά το θέμα είναι, θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε τις προτάσεις πριν από τις ευρωεκλογέ. Εμείς είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Μπορούμε και τα δύο χρονικά παράθυρα να σεβαστούμε. Αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν επιλογές οι οποίες θα μας οδηγήσουν προς τη μία ή την άλλη λύση. Και αυτό θα το ορίσετε εσείς. Την ε, προηγούμενη φορά, το Δεκέμβριο του 2013, ήμασταν, ε, είχαμε αποφασίσει και έτσι είχε χαθεί τελείως ένα έτος γιατί καθυστερήσαμε στην υλοποίηση και μέσα σε ε, εποχές δύσκολες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε ένα ολόκληρο χρόνο. Βρεθήκαμε δηλαδή λίγο πολύ στα μισά του πολιτικού δημοσιονομικού ε, σχεδίου να αρχίσουμε να, υλοποιούν, να υλοποιούμε. Εάν όμως θέλουμε τα επενδυτικά μας προγράμματα ε, είτε πρόκειται για την οικονομική ανάκαμψη, για το εργατικό δυναμικό, για τη βιομηχανία, να υλοποιηθούν, τότε δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο. Έχουμε ήδη καθυστέρηση 2019, 2020, 2020, 2022. Και εδώ το τωρινό πολιτές δημοσιονομικό σχέδιο θα καθυστερήσει να εγκριθεί, να υλοποιηθεί μάλλον. Θα κινδυνεύουμε να δούμε περικοπές και όποιος θέλει να υπηρετήσει την Ευρώπη, όποιο θέλει από το 1η Ιανουαρίου του 2021 είναι έτοιμο για δράση, πρέπει πιο νωρί να έχει κάνει τη δουλειά του, να είναι προετοιμασμένο, και αυτό είναι το δίδαγμα το οποίο αποκομίζουμε από τι τελευταίες διαπραγματεύσει του πολιτή δημοσιονομικό σχεδιασμό μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και στον επόμενο χρόνο είμαι στη διάθεσή σα και περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλε τι προτάσει σα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την πάρα πολύ αναζωογονητική, διεγερτική θα τη χαρακτήριζα συναρπαστική αυτή ομιλία. Καλέσατε όλους μας να αναλάβουμε πλήρως τις ευθύνες μας. Α, πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε από την Ευρώπη και τι περιμένουμε από την Ευρώπη και πρέπει γι' αυτό βέβαια να καταρτήσουμε έναν προϋπολισμό που να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και ο οποίος να μπορεί να είναι βιώσιμος. Θα ξεκινήσει λοιπόν τώρα η συζήτηση. Γνωρίζω ότι θα πρέπει σε λιγότερο από μία ώρα να διακόψουμε, οπότε θα παρακαλέσω όλους ε, όσους λάβουν το λόγο να είναι στο δυνατόν ε, πιο συνοπτικοί. Δύο λεπτά θα έλεγα να έχει ο καθένα ως χρόνο αγόρευση και αν τον τηρήσει θα είμαι ευγνώμονα. Καταρχάς θα ακούσουμε του ε, εισηγητέ ε, για το πολιτέ δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Η κυρία Τομά, η κυρία Σόλμπριχτ, ποιο θέλει πρώτο το λόγο. Μην το κουράσετε μεταξύ σα, ποιο θα αποφασίσει ο κύριο Σόλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Νομίζω ότι είναι ένα έγγραφο το οποίο το περιμέναμε, σας ακούσαμε και πριν ε, από αυτό το έγγραφο που κάνατε κάποια παρουσίαση. Είχαμε ε, λάβει κάποια γνώση για προπαρασκευαστικές ενέργειες και τώρα έχουμε πλέον το τελικό αποτέλεσμα ενώπιον μας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο, διότι πρόκειται για κάτι καινούριο στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται εν γέννη τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι μια προσπάθεια, κατά την άποψή μου, αλλαγής μεθοδολογίας μια προσπάθεια να είστε πολύ πιο συγκεκριμένοι στις εργασίες σας. Και πράγματι το θέμα είναι αυτό ακριβώς, να συζητήσουμε συγκεκριμένα και για συγκεκριμένα ζητήματα. Γι' αυτό και το θέμα δεν είναι μόνο η ανάλυση του κόστους, πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά, αλλά και το θέμα της προστιθέμενης αξίας. Και νομίζω ότι το εξηγήσατε με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και έτσι ακριβώς πρέπει να εννοήσουμε την προστιθέμενη αξία. Μην ξεκινήσουμε επιστημονική συζήτηση για το τι εστί προστιθέμενη αξία, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί μια τέτοια συζήτηση. Αυτό επίσης που είναι άκρος ενδιαφέρον είναι το τελευταίο τμήμα, τα σενάρια δηλαδή. Ποιες θα είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτινόμενων σενάριων. Για μας φυσικά και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί μας δίνει τροφή για σκέψη αυτό είναι το υλικό που έχουμε μπροστά μας για να δούμε ποιε θα είναι οι πιθανέ επιπτώσεις. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι το εξή. Αν δούμε αναλυτικά τα διάφορα σενάρια και τις δικές σας προτάσεις, ε, βλέπουμε ότι ανάλογα με το σενάριο διαφορετική είναι και απαιτούμενη προσέγγιση, διαφορετικές είναι οι μέθοδοι και διαφορετικά θα πρέπει να ε, θεσπιστούν και οι πολιτικές, δηλαδή αυτό που εσείς περιγράφετε στα σενάρια. Είναι η αλλαγή των ε, πολιτικών. Μιλάμε για αλλαγή στην πολιτική, τη γεωργική ή την πολιτική συνοχή. Δεν μιλάμε μόνο για τους οικονομικούς πόρους, για τα κονδύλια. Το έγγραφο δεν αφορά μόνο τον προϋπολισμό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θέλουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι η συζήτηση, έτσι τίθεται πλέον η συζήτηση, μέσω μεν του προπολογισμού, αλλά υπερβαίνοντας ουσιαστικά τα αυστηρά δημοσιονομικά ζητήματα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά θέλω να σα κάνω μια ερώτηση για τη διαδικασία. Αν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει συγκεκριμένε πολιτικέ και προτάσει από τι διάφορε δικέ μα κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, θα πρέπει να έχουμε και κάποια αφετηρία γι' αυτό. Και το ερώτημά μου είναι, χρειάζεται πολιτική απόφαση για το σενάριο ή ας το πούμε για το μοντέλο. Εσείς θα μου απαντήσετε αν θεωρείτε ότι ναι ή όχι. Δηλαδή, Συμβούλιο, Κομισιόν, Κοινοβούλιο. Πρέπει να έχουμε λάβει μια πολιτική απόφαση καταρχάς για το τι θέλουμε και μετά να περάσουμε στη συζήτηση πάνω στα σενάρια και τα διάφορα στοιχεία τους. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα η πολιτική απόφαση ή η δική σας νομική πρόταση που θα κατατεθεί σε αρχές του επόμενου έτους, στο πρώτο εξάμεινο, θα είναι η πρόταση για την απόφαση. Δηλαδή, για να το επαναλάβω, ή θα έχουμε την απόφαση πριν την νομοθετική πρόταση που θα είναι με τα απόρρια της απόφασης ή η πρότασή σας θα προηγηθεί της απόφασης. Από πολιτικής πλευράς είναι λεπτό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν θέλουμε να εργαστούν οι επιτροπές μας έχουν εντελώ διαφορετικές ιδέες για τις διάφορες πολιτικές και δεν μπορούν να επεξεργαστούν τα διάφορα σενάρια και τις διαφορετικές ε, πολιτικές. Πρέπει κάπου να εστιάσουμε. Γιατί αλλιώ θα είναι απλά μια δονητική άσκηση χωρί κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ερώτηση προ εσά. Ευχαριστώ κυρία Τωμά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον Επίτροπο. Βέβαια, μόλις έλαβα το έγγραφο και δεν είχα το χρόνο να το διαβάσω. Ήδη από τώρα όμως θέλω να χαιρετήσω την προσέγγιση που προτείνεται, η οποία ε, δείχνει ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επίσης, μας δίνει πολύ ενδιαφέρουσες πίστες για το που πρέπει να πάμε και για μια ακόμη φορά δείξατε τη διάθεσή σας για διάλογο. Βέβαια, σήμερα, αυτό που κάνετε εσείς είναι ότι κηρύστε την έναρξη αυτού του διαλόγου για το μέλλον της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί δείξατε ιδιαίτερα ε, διάβγεια περιγράφοντας την κατάσταση. Μιλήσατε για τις εκπτώσεις ιδίους πόρους, ε, τη... τα δημοσιονομικά, την προσθέμενη αξία. Είπατε επίσης ότι ο προϋπολογισμός ε, δεν έρεται στο ύψος των προσδοκιών που πρέπει να εκπληρώνει ο προϋπολογισμός. Και πράγματι το ζήσαμε, το είδαμε και με την αναθεώρηση του πολίτου του πλαίσιου και θέλω εδώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχία στην οποία όλοι συνεισφέραμε και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό. Όμως το είδαμε στην προκειμένη περίπτωση, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ελλειπής χρηματοδότηση που έχει προσλάβει δομικό χαρακτήρα, το είπατε και εσείς. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Αντίθετα τώρα, είπα μέχρι στιγμής που συμφωνώ μαζί σας και περνάω στην άλλη όψη του νομίσματος. Αντίθετα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τη συζήτηση αυτή, έχουμε κατά την άποψή ένα πρόβλημα. Το πρώτο στοιχείο του προβλήματος είναι ότι έχουμε μία ημερομηνία ε, που την προβλέπει ε, το Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για το μελλοντικό πολιετές η Κομισιόν. Πριν την 1η Ιουλίου του 2018 είναι αυτή η προθεσμία και είναι καταγεγραμμένη. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί, απλά ήθελα να το υπενθυμίσω. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του συμπεράσματος στο οποίο καταλήγεται δεν έχουμε πολύ χρόνο και επιθυμείτε να έχουμε ολοκληρώσει στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και νομίζω σωστά είπατε ότι πριν τα τέλη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου πρέπει τουλάχιστον να έχουμε καταλήξει σε, στην ολοκλήρωση της πρώτης έστω συζήτησης για το επόμενο πολιετές μετά το 2020, αλλά απ' την άλλη μας ταυτόχρονα να περιμένουμε. Αυτή την αντίφαση θα ήθελα να την υπογραμμίσω. Λαμβάνοντας ιδέως υπόψη, όπως είπε ο συνάδελφος και συνεισηγητής, επικρατεί κάποια σύγχυση, διότι ξεκινά μια συζήτηση για το χρηματοοικονομικό μέλλον, το δημοσιονομικό μέλλον της Ένωσης, χωρίς καμία στρατηγική μέχρι στιγμής να έχει χαραχθεί. Και ο προπολογισμό προηγείται τη στρατηγικής και από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, είναι συχνό το φαινόμενο. Αλλά αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Δυσχεραίνει τη θέση μας. Είχαμε τη στρατηγική 2020 και σε αυτήν προσαρμόσαμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2014-2020. Τώρα τα πράγματα περιπλέκονται. Παρ' όλα αυτά, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και επειδή δείχνει εδώ το ρολόι ότι μακρηγόρησα και ανάβει το κόκκινο φωτάκι και σε το συγγνώμη γι' αυτό. Τέλος πάντων, η ερώτησή μου και έρχομαι σε αυτήν είναι θα πρέπει να κινηθούμε ε, συντονισμένα και παράλληλα σε ό,τι αφορά και τα θέματα της στρατικής και στα θέματα τα δημοσιονομικά. Αλλιώς δεν θα ε, καταφέρουμε να είμαστε πιστοί στο ραντεβού που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τέλη της κοινωνικής περίοδου το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το 2000, μετά το 2020. Να γνωρίζετε ότι η δική μου ομάδα είναι δετεθειμένη να εργαστεί, από κοινού με Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Από κοινού μαζί τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Και να έχουμε αυτό το διάλογο που εσείς ε, εγκαινιάσατε σήμερα και για το οποίο θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα είμαστε εργάσιμοι, αλλά θα είμαστε και απαιτητικοί. Σας ευχαριστώ κύριε Τωμά. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο εισηγητές των ιδίων πόρων, αλλά τους θέρμο παρακαλώ να μην ξεπεράσουν το δίλεπτο. Θα ήμουν ευγνώμων γι' αυτό. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, διαμαρτύρομαι για την κακή μεταχείριση. Όχι πλάκα κάνω. Κύριε Επίτροπε, Ε, όχι. Πρέπει να διασκεδάσετε αυτέ τι αμφιβολίες. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο ευγενικό γίνεται. Καλά, ας περάσουμε στου ιδίους πόρου καλύτερα, για να δείξω ότι πολλά από αυτά που μα είπε ο επίτροπο δυστυχώ δεν μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά. Ε, συγχαρητήρια για την ομιλία σα. Καταρχήν, να σμηδενίσουμε το χρονόμετρο. Εντάξει, έχετε μισό λεπτό επιπλέον. Κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια για τη μαχητικότητα, ε, και το, την ομιλία σας. Και είστε και πολύ επιδέξιος και ικανός κατά τη γνώμη μου, γιατί μας κάνατε μια σκιαγράφηση της κατάστασης για να μας βοηθήσετε να περιμένουμε ουσιαστικά, να κάνουμε υπομονή. Γιατί μας λέτε αυτά θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν γίνεται από τώρα, γι' αυτό θέλουμε λίγο χρόνο για να το πραγματοποιήσουμε. Δείξτε υπομονή. Ε, όλους παραδόξως θεωρώ ότι είναι αρκετά συνετή αυτή η στάση. Πρώτον, γιατί στο μέτρο που δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του Brexit και τι δημοσιονομικέ επιπτώσει, πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε. Οι Βρετανοί, λέει, ε, θα οφείλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 60 δισεκατομμύρια. Αν το δεχτούν αυτό το ποσό και το πληρώνουν κάθε χρόνο 10 δισεκατομμύρια το χρόνο για 6 χρόνια, δεν θα έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα. Θα πρέπει όμω να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποια θα είναι η έκβαση του Brexit και αν θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση ε, κάποιων πολιτικών. Βέβαια βλέπω να διαφωνεί η Σαμπέλ Τωμά, εγώ πάντως εμένω και επισήμω στη θέση μου και την επιβεβαιώνω. Σε ό,τι αφορά επίσης ε, τη χρηματοδότηση σε περίπτωση που δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Είστε αρκετά αισιόδοξο όταν λέτε ότι θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις ε, εισφορές τους με βάση το ΑΕΕ. Ε, κοινό από την υπόθεση ότι για πολλούς καθαρούς εισφορείς η ιδέα της αύξησης ε, της εισφοράς για να μειωθεί η μείωση της ε, συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού του Ηνωμένου Βασιλείου είναι όνειρο θερινής νυκτός. Και φαντάζομαι για τους ιδίους πόρους θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ιδίους πόρους που θα επιβαρύνουν άμεσα τους πολίτες αν αυξηθεί η τιμή του α ή του β προϊόντος για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή υπεραξία, όχι, δεν νομίζω ότι να περάσει αυτό το επιχείρημα. Αλλά το θέμα των ιδίων πόρων αποκτά κέρια σημασία, νευραλγική. Και νομίζω και αυτό μας ζητήσατε, να ακολουθήσουμε τη λογική της έκθεσης Μόντι. Όμως ε, η έκθεση Μόντι έχει δύο άξονες και εσείς μιλήσατε μόνο για τον ένα, την COP21 και τις συνέπειες στην ενέργεια και την προστασία του κλίματος. Υπάρχει όμως και ένας άλλος άξονας, ισότιμος, ε, να γίνει πιο σωστή και πιο δική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και εκεί έχουμε πόρους που αφορούν την εναρμόνιση του φόρου για τις εταιρείε, επίσης εναρμόνιση του συντελεστή ΦΠΑ ε, και εισφορά κάποιου ποσοστού. Αυτά έχουν νόημα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καλάθι δύο πόρων που θα συμβάλλει ε, και θα ικανοποιεί και αυτές τις δύο αυτές οι δύο κατευθύνσεις, αυτούς τους δύο άξονες. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ για το έγγραφο προβληματισμού, κύριε Επίτροπε. Ο προβληματισμός μου, για τον προβληματισμό σας θα είναι πολύ σύντομος. Εγώ απλώς ε, θα περιοριστώ στο να ακούσω σήμερα το απόγευμα και ε, η δικαιολόγηση ότι δεν είναι και πολύ πλούσιο το έγγραφο προβληματισμού και όχι πολύ ακριβές για το θέμα των ε, εσόδων ισχύει, αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι θα βάλετε τα δυνατά σας και έχετε το κουράγιο να προσπαθήσετε ε, να προτείνετε νέους ιδίους πόρους. Ίσως αξιοποιώντας το Brexit ως ε, παράθυρο ευκαιρίας και την έκθεση Μόντι ως βάση. Δεν ε, αναφέρεται πουθενά στο έγγραφο ότι θέλετε να καταργήσετε όλες τις επιστροφές, στα rebate. Ε, αυτό είναι αρκετά αισιόδοξο, που είπατε ότι θέλετε να τα καταργήσετε αυτά τις επιστροφές, αλλά έχουμε και την αρχή του φωτενευλό. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των ε, εξόδων. Αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Και πέρυσι προσπαθήσαμε να καταργήσουμε τις επιστροφές, τα rebates, αλλά για μερικές χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένες και της Γερμανίας, Ζητήσαμε αποζημιώσει ε, φάπαξ κατά αποκοπή ποσού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσουμε μια δίκαιη θέση μέσα το, μέσω των δαπανών του προπολογισμού. Αυτά προ το παρόν, υπακούοντα και στην έκκληση του Προέδρου να είμαστε λακωνικοί. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στους συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών και να με συμπαθάτε, αλλά θα σας επιβάλλω το δίλεπτο ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Ξέρω όμως ότι είστε υποδηματικός συντηρήση του χρόνου. Ευχαριστώ. Ε, μην αρχίζετε ακόμη το χρονόμετρο. Εντάξει, θα έχετε ακόμη πέντε δευτερόλεπτα. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ε, παρουσίαση του εγγράφου και την ε, αφοσίωσή του και τη στράτευσή του στο θέμα αυτό. Θα είμαι λακωνικός, τηλεγραφικός. Θεωρώ ότι είναι θετική μια συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για λόγους προβλέψιμότητα, όπω είπατε, και μάλιστα καλό θα ήταν αυτό να γίνει ε, τρέχουσα στις ε, ε, κοινοβουλευτικές θητείες πριν τι επόμενε ευρωεκλογέ. Και σημαντικό είναι να έχουμε κατά τη θητεία αυτή τη συμφωνία και υπάρχει καλή διάθεση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω και το Συμβούλιο να δείξει την ίδια προθυμία και να επισπεύσει τα πράγματα. Ε, έχουμε τη στρατηγική του 2020 ε, μιλάει για την απασχόληση, τι κλιματικέ αλλαγέ την καταπολέμηση τη φτώχειας, εξάλληψη τη φτώχεια, ε, παιδεία, επενδύσεις στην ανάπτυξη. Έχουμε βέβαια άλλη προτεραιότητα τώρα, την ε, ασφάλεια και την άμυνα. Περιμένουμε και τι συνέπειε του Brexit. Ναι, αν περιμένουμε όμω πολύ για να ολοκληρωθούν οι συνέπειε, κινδυνεύουμε να μην έχουμε επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί οι τελικέ επιπτώσει του Brexit δεν ξέρουμε πότε θα διαμορφωθούν. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε εμεί να προχωρήσουμε στο έργο μα. Και ξέρω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να περικόψει τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, υπάρχουν προτεραιότητες που δίνονται και οφείλουν να ενισχυθούν. Και αυτό που είναι σαφές κατά τη γνώμη μου είναι ότι, χρειαζόμαστε, είναι ότι έχουμε μια στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Ευρώπη 2020 όμως στρατηγική παρατεταμένη στο χρόνο και με νέες προτεραιότητες προϋποθέτει αύξηση της, του ποσοστού του ακαθάριστου εχώριου εισοδήματος για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ναι, μεν περισσότερη ελαστικότητα, αλλά θέλουμε και καλύτερη προβλεψιμο... προβλεψιμότητα και, και να έχουμε μέγιστη ελαστικότητα θα χρειαζόμασταν ένα χρόνο μόνο σχεδιασμός. Αλλά δεν αρκεί αυτό για την προβλεψιμότητα. Μας μίλησατε για 5 συν 5. Τι ακριβώς εννοείται. Θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί μόνο με μία πενταετία δεν έχουμε επαρκή προβλεψιμότητα. Επίσης, τι θα γίνει με την εκτέλεση στην πολιτική συνοχής. Ακόμη δεν έχουν ορίσει όλα τα κράτη-μέλη τους διαχειριστικούς τους φορείς, τις διαχειριστικές αρχές για την πολιτική συνοχής. Επίσης, η αιρεσιμότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις επιχειρήσεις, στους φοιτητές, στους πολίτες, στους ερευνητές, στις περιφέρειες. Γιατί η αιρεσιμότητα το πολύ μπορεί να εφαρμοστεί και να ισχύσει για τα κράτη-μέλη. Ποτέ όμως για τα κονδύλια και τα προγράμματα. Ε, μιλήσατε για προστιθέμενη αξία, για υπεραξία. Αυτό όμως προϋποθέτει μια πολιτική στάθμιση και επιπλέον θα πρέπει να εξετάσουμε το κόστος της μη ύπαρξης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Γιατί πριν απο 34 χρόνια κανένας δεν θεωρούσε ως υπεραξία ή προστιθέμενη αξία όλη την εξωτερική ενίσχυση που παρέχουμε με, όλα τα μηχα... με όλους τους μηχανισμούς και τα μέσα που χρειάστηκε να ενισχύσουμε ε, μέσω γειτονίας ή αντιμετώπιση της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης. Αυτά ευχαριστώ. Η κυρία Γκουάρτια Θάμπαλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο Έτιγκερ. Εγώ θα κάνω το αντίστροφο από την Ιζαμπέλη. Θα ξεκινήσω δηλαδή με τι δεν μου αρέσει και θα ολοκληρώσω με τα θετικά. Έχω ένα ζήτημα αρχής αλλά και στρατηγικής με αυτό το reflection paper της Κομισιόν, διότι νομίζω ότι ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα λαβύρινθο, ε, συζήτηση λαβύρινθόδη για διάφορα σενάρια. Αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ευρώπη και θέλουν να τερματίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμα, ε, εργάζονται αόκνος προς αυτό το σκοπό. Και εμεί, ως Ευρωπαίοι και φιλοευρωπαίες δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε προς το μέλλον ή να δρούμε χωρίς να σκεφτόμαστε σκεφτούμε προηγουμένως. Αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Ε, το προ-Brexit δημοψήφισμα, μετά Brexit και άλλος ένας χρόνος προβληματισμού και να συζητούμε χωρίς να βρούμε διότι ο κόσμο που πιστεύει στην Ευρώπη έχει απογοητευτεί γιατί δεν βλέπει αντίδραση εκ μέρου μα. Δεν βλέπει να τα αποκρινόμαστε στα άμεσα προβλήματα των συμπολιτών μα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θέλουμε είναι γνωστό. Το ξέρουμε πολύ καλά. Και όταν συζητήσουμε με το πολιετέ δημοσιονομικό και το βλέπω όταν μιλούμε στις, για τα θέματα αυτά στι ειδικέ επιτροπέ, για τη γεωργία, την εξωτερική πολιτική ανάπτυξη, γεωργία κτλ. Όταν ζητάμε του αδελφούς να μα πούν τι θέλουν για το επόμενο πολιετέ, δεν μα λέει κανεί καθίστε να δούμε πρώτα τι σενάριο θα επιλέξουμε απαντούν. Ε, στην Ήτρε θέλουμε πιο πολλά χρήματα για τον το 2020, να συνεχίσει να λειτουργεί το πρόγραμμα COSME, να υπάρχουν επενδυτικά σχέδια. Από την Επιτροπή Γεωργίας μας λέει να μεταρρυθμιστεί η ΚΑΠ χωρίς όμως περικοπές των κονδυλίων. Οι της συνοχής μας λένε θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εδαφική συνοχή της Ευρώπης. Άρα τα λένε όλοι ξεκάθαρα και κανένας δεν μας λέει θα εξαρτηθεί από το ποιο σενάριο θα επικρατήσει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα ε, και νομίζω επειδή μας ζητήσατε υπομονή, αρκετή υπομονή έχουμε κάνει. Ε, δεν μιλώ βέβαια συγκεκριμένα για το έγγραφο, μιλάω γιατί υπήρξε κάποια αμφίσιμη στάση της Κομισιόν μέχρι τώρα. Και έρχομαι τηλεγραφικά στα θετικά πολύ καλό να σταματήσουμε τα τσεκ, επιστροφές, εκτόσεις. Ε, καλό να συμπεριληφθούν όλα τα κονδύλια, όλα τα ταμεία που είναι εκτός περιπολισμού, να μπουν στον περιπολισμό. Και πολύ καλό τέλος που ξεκινάει η συζήτηση για τους ίδιους πόρους ε, με συγκεκριμένες ιδέες, προτάσεις και ακόμη ε, κάτι καλό που μπήκε στο τραπέζι το θέμα της διάρκειας. Πρέπει να συζητήσουμε το είδος του πλησίου, αλλά το 5 συν 5 Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που ισορροπεί τι ανάγκε μεταξύ ευελιξία αφενό και προβλεψιμότητα αφεντέρου. Τέλο, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για τον συμβιβασμό και για την, μάλλον για τη δέσμευσή σα ότι θα συμμετέχει σε αυτέ τι διαδικασίε στο Κοινοβούλιο και αυτό συνιστά ουσιαστική αλλαγή. Γιατί έχει γίνει σημαντική δουλειά ε, και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να βοηθούμε εμεί από το Κοινοβούλιο με τι επιτροπέ τη διάφορε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κέλμελ που όμως δεν είναι μέσα στην αίθουσα από ό,τι βλέπω. Άρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπχέ. Όχι ως εισηγητή πια για τους ίδιους πόρους, αλλά ως συντονιστή της ομάδος Άλντε. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, αν μου επιτρέπετε. Ή στον επόμενο μιλτή, ή στον ε, έναν από τους εξευωνίμων ή εκδεξιών καθήμενο συνάδελφο. Ναι, εσείς δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και για τον κύριο Επιτρόπο που ήρθε εδώ. Δύο ερωτήσεις και κάποια σχόλια από πλευρά μου. Κύριε Έτιγκερ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για τους ορυφωσικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς ε, αντιμετώπισης κρίσεων. το ποσό που διατίθεται, πόσο, ε, σε ποιο ποσοστό του προπολογισμού το κράτο μελών ανέρχεται. Θα έλεγα γύρω στο 1% και σε ό,τι αφορά τι δικέ μα δαπάνε, σε σχέση με τι δαπάνε στο δημόσιο τομέα των ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σφίγγει το ζωνάρι. Τα κράτη-μέλη επίσης έχουν σφίξει το ζωνάρι, τα περισσότερα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο από τα κράτη-μέλη τελικά. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους και τις προτάσεις Μόντι και τη μείωση ε, των εισφορών των κρατών μελών. Μάλιστα, να το δούμε. Ο προπολογισμό της Ένωσης δεν πρέπει να αυξηθεί αν μου Πρόεδρος, θα ήθελα να μιλήσω για την κοινή πολιτική. Έχω ακούσει κάποιες φήμες ότι θα περικοπούν τα κονδύλια και με ανησυχεί αυτό γιατί θέλουμε να παράγουμε τρόφιμα για τους Ευρωπαίους και η γεωργική παραγωγή είναι επίσης πολύ σημαντικός ε, φορέας ε, ε, σε ό,τι αφορά και την κλιματική αλλαγή. Όταν απαιτούμε από αυτούς περισσότερες προσπάθειες σε αυτό το μέτωπο, δεν είναι και λογικό να μειώνουμε την υποστήριξη που τους παρέχουμε. Ήμουν σύντομη, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τάχο. Τάραντ μάλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, πολύ ε, δυναμική και ξεκάθαρη παρουσίαση των προθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας υπόσχομαι ότι οι πράσινοι θα συζητήσουν ε, πολύ θερμά αυτά, αυτές τις ιδέες και θα υποβάλουν ως συνήθως τις επικοδομητικές προτάσεις. Τρεις ε, σύντομες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι το θέμα των ιδίων πόρων είναι πολύ σημαντικό. Και αν εμείς υπό τη δική ε, σας ηγετικό ρόλο επιτύχουμε κάτι για τους ιδίους πόρους θα είναι ιστορική στιγμή, όπως θα έλεγε ένα ιστορικό σαν και Και αν θέλετε υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητήστε την ελεύθερα, μην τρέπεστε, γιατί δεν θέλουν όλα τα κράτη-μέλη κάτι τέτοιο. Επίση, κανεί δεν μπορεί να. Το, το πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατο. Ο πατέρα μου ε, ήταν επιστήμονα, ε, παρακολουθούσε ε, τα θέματα ε, διαμόρφωση του κλίματο. Οπότε το θέμα των κλιματικών αλλαγών με αγγίζει ιδιαίτερα και την ομάδα μου. Επίση, το θέμα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε επταετία. Ξέρουμε ότι ο συγκεκριτή μα, ο, ο κύριο Μουρεσάν, προτείνει πενταετία. Εσεί είπατε πέντε συν 5 ίσως θα μπορούσαμε να το συνδυάσουμε ή να το σχετίσουμε με την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάρκεια της από το να ερχόμαστε εδώ και να βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι ευρωβουλευτές είχαν λάβει την απόφαση και δεν επιδέχεται αλλαγέ. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να σπάσουμε τον πάγο και πραγματικά θα ήταν ευχή έργων αν τα καταφέρουμε. Ίσως να ακούγεται ως προσβολή, κακός, παρα, άστοχος παραλληλισμός, αλλά στη Σοβιετική Ένωση είχαμε το 5 5 και μόνο Χρουσόφ είχε αυτά, αλλά πέτυχε. Συγγνώμη. Μάλιστα, ο κύριος ε, Αρνότ. Όχι, απουσιάζει. Οπότε η κυρία Νιριάντα. Όχι. Σόλτεκ. Δεν τους ευχαριστώ για τη λακωνικότητά τους. Μόνικα Χολμάιερ. Εγώ είμαι εδώ. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω καταρχάς ότι μου φαίνεται πολύ θετικό το γεγονός ότι παρουσιάζει εδώ ένα έγγραφο ε, με ανοιχτή διατύπωση, όχι ένα έγγραφο στο οποίο δηλαδή έχουν παγιωθεί όλες οι πιθανές θέσεις. Είναι πολύ καλό να γίνει αυτή η συζήτηση, ιδιαίτερα του τι σημαίνει Ευρώπη, τι προσφέρει επιπλέον ως υπεραξία η Ευρώπη, χωρί να χρειάζεται να εμβαθύνουμε ιδιαίτερως. Νομίζω ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε κάποιες θέσεις από αυτές τις οποίες έχουμε συνηθίσει να παραλαμβάνουμε και οι οποίες δεν είναι απαραίτητα πάντοτε χρήσιμες. Η αρχή μιας περίοδου 5 συν 5 ετών είναι χρήσιμη, γιατί ξεκινάμε κάθε πενταετία να συζητούμε εάν χρειάζεται μια εκ των θεμελίων τροποποίηση των ε, προγραμμάτων μας σε κάθε αρχή πενταετίας. Βεβαίως είναι καλό κανείς να έχει ανοιχτό πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει κάθε φορά να συζητούμε για μια νέα μεταρρύθμιση η οποία θα τεθεί σε ισχύ δύο χρόνια αργότερα, γιατί νωρίτερα δεν μπορούν να την υλοποιήσουν οι εθνικές νομοθετικές αρχές και ούτως ή άλλως καθυστερεί ακόμη περισσότερο η πραγματική της εφαρμογής στην πράξη. Η πραγματικη της εφαρμογη στην πραξη η πενταετια συν μια ενδιάμεση αναθεώρηση και άλλη μια πενταετία στη συνέχεια είναι πολύ πιο ε, χρήσιμη ως λύση. Ε, επίσης, σε θέματα που έχουν να κάνουν ε, με ε, προβληματισμό, θα ήταν καλό να ξανασκεφτούν τα κράτη-μέλη ποιες υπηρεσίες είναι πράγματι απαραίτητες για το μέλλον της Ευρώπης, ποιες ενδεχομένως θα μπορούσαν είτε να περισταλούν στην έκτασή τους, είτε και να καταργηθούν. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Υπάρχουν τομεί επίση όπω ο τομέα τη γεωργία, όπου διαρκώ ακούγεται, ε, διαρκώς γίνεται λόγο για την επανεθνικοποίηση. Ε, να επιστρέψει δηλαδή στι εθνικέ αρμοδιότητε, ε, τότε ίσω θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τι σχετικέ ευθύνε και όχι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό, γιατί με συγχωρείτε, αλλά όταν γίνονται τόσε επανεθνικοποίησει, τόση συζήτηση μάλλον για επανεθνικοποίηση, γιατί θα πρέπει να τα πληρώνει αυτή την επανεθνικοποίηση και τη σχετική πολιτική ο ευρωπαϊκό προπολογισμό, α ορίσουν τα κράτη-μέλη τι δικέ του προτεραιότητε. Και μάλιστα στον τομέα τη γεωργία. δεν είναι πάντα τόσο αυτονόητο, θα το πω έτσι, μια μεγάλη βιομηχανική επιχείρηση να λαμβάνει επιδότηση σημαντική από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό παρότι είναι πλήρως ανταγωνιστική. Ενώ σε άλλους τομείς που έχουμε ανταγωνιστικό έλλειμμα, όπως η παραδείγματι στην γεωργία, που πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα ή να ορίσουμε ποιοι είναι οι όροι για τους οποίους την ε, ε, την υποστηρίζουμε, γιατί βεβαίω εγώ είμαι υπέρ της παραγωγής των τροφίμων στην Ευρώπη και υπέρ της ενίσχυσης της γεωργικής ε, παραγωγής όπου υπάρχει ανάγκη, αλλά θα ήταν καλό να κοιτάξουμε πού υπάρχει ανάγκη. Και επίσης ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πού πραγματικά χρειάζονται τα χρήματα για την καινοτομία και την έρευνα, γιατί εκεί, από εκεί μάλλον θα κρυθεί και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για να έχουμε καινοτομίε που θα μπορούμε να προσφέρουμε στον πολίτη για το μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Γκάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολύ έπαινοι για το έγγραφο προβληματισμού. Θα τους επαναλάβω κι εγώ. Θα δώσω έτσι και την ευκαιρία σε κάποιους συναδέλφους, χαίρετε, να λάβω το λόγο, να λάβουν το λόγο. Εγώ θα επικεντρωθώ όμως περισσότερο στα θέματα που έχω κάποιες επικρίσεις να διατυπώσω. Θα περίμενα, την Τίνκερ, περισσότερη παρησία στο θέμα των ιδίων πόρων. Γιατί η έκθεση Μόντι κάνει εννέα προτάσεις. Κάποιοι είπαν εννέα προτάσεις, θα οδηγήσουν σε μια αναδιατύπωση από το Συμβούλιο που θα μετατραπεί σε δικαιολογία του γιατί δεν μπορεί να υλοποιηθεί τίποτα από αυτά και ίσως θα ήταν καλύτερο, είναι πιο δυναμική η πρόταση και πιο θαραλέα η πρόταση της ομάδας του Μόντι. Και τώρα από τις 9, αν καταλαβαίνω καλά, επιλέγετε τις δύο. Αλλά θα έλεγα ότι στα γερμανικά, όπως τα είπατε, ήταν μάλλον διστακτική διατύπωσή σας. Εγώ επιμένω ότι πρόκειται για μια σημαντική συμβολή, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημαντική υποχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που καθίσατε σαφής, χρόνο με το χρόνο, και γι' αυτό ήρθε η ώρα να πούμε με θάρρος αυτές τις προτάσεις θέλουμε να κάνουμε και έτσι προχωρούμε. Μια δεύτερη επισήμανση που φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και πολλούς αδελφούς από την περιφερειακή πολιτική είναι η εξή. Ότι όντω έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να γίνει συζήτηση για μετατόπιση κονδυλίων. Να την κοιτάξουμε, να την εξετάσουμε. Βεβαίω. Πρέπει να κοιτάξουμε και ποια είναι τα ποσοστά απορρόφηση, ποια είναι η θέση τη πολιτική συνοχή που δεν είναι η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θα έκανα το παν για να υπερασπιστώ την πολιτική της συνοχής, όπως έχει. Τα δε σενάρια τα οποία ακούγουμε να περιγράφονται τείνουν να δείχνουν ότι η πολιτική συνοχής, ναι, μπορεί να είναι η, η απεικόνηση πιστή, δεν είναι τα πάντα τέλεια στην πολιτική συνοχής, αλλά η πολιτική συνοχή σε κάθε τομέα και σε κάθε περιφέρεια μπορεί να προσφέρει τεράστια υπηρεσία στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε, στο πιο κοντινό επίπεδο σε αυτούς για να συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ τον Επίτροπο Έτιγκερ για την παρουσίαση και το έγγραφο προβληματισμού που υπέβαλε. Είναι πολύ επίκαιρο, κατά τη γνώμη μου, το έγγραφο αυτό. Και όπως είπατε κι εσείς, ο χρόνος πιέζει, κύριε Επίτροπε. Έχουμε αυτή τη στιγμή την ε, αξιολόγηση αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να εγγύψουμε στο μελλοντικό, στο επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση αποκλείεται να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές και τις προτεραιότητές μας. Χωρίς χρήματα και χωρίς κονδύλια, χωρίς χρηματοδότηση, αποκλείεται να ε, καταλήξουμε σε σωστές προτεραιότητες και να χαράξουμε μια σωστή κατεύθυνση για την ανάπτυξή μας. Τώρα φυσικά βρισκόμαστε στην ε, αρχή της συζήτησης, ε, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε δεδομένες και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε. Δεν θα πρέπει να ξεκινάμε τα βασικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το κύριο θεμέλιο είναι η αλληλεγγύη. Βέβαια, δεν είναι το μοναδικό θεμέλιο, γιατί ας μην ξεχνούμε, είμαστε μέλη τη Επιτροπής Προϋπολογισμών. Αλλά θέλουμε έναν προϋπολογισμό που θα ε, προσανατολίζεται στην ε, υλοποίηση αποτελεσμάτων. Ένα τέτοιο προπολογισμό ε, θα πρέπει να είναι και ο προπολογισμό του 2018. Επίσης, ε, έχουμε το επενδυτικό σχέδιο Juncker και τα σχέδια του επενδυτικού αυτού σχεδίου θα έχουν προστιθέμενη αξία γιατί θα εμπλέξουν ε, χώρες και περιφέρειες, οπότε σαφώς θα έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και γι' αυτό θα είμαστε υπόλογοι και εμείς. Κατά την προετοιμασία του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που θα καλύπτει μία περίοδο μετά το 2020. Έχω μία ερώτηση. Είπατε ότι το επόμενο α, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να έχει μία διάρκεια 5 συν 5 έτη. Κανένα πρόβλημα. Ποιες όμως είναι η προσδοκία σας για την επόμενη δεκαετία. Για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, για παράδειγμα. Γιατί είχαμε αυτή τη στρατηγική μέχρι το 2020. Έχουμε ετοιμάσει μια νέα στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Γιατί ίσως και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη κατά την προετοιμασία των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Και για το Brexit, μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων. Και πιστεύω ότι το θέμα συνδέεται και με το επόμενο ΔΕΛΤΑΠΗ. Μετά το Brexit λοιπόν θα έχουμε υποχρηματοδότηση. Οπότε, αν δεν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις μας και οι εκτιμήσεις μας και δεδομένων των νέων προκλήσεων όπως είναι η μετανάστευση, η ασφάλεια και ούτω καθεξής, μήπως θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και πώς αυτό θα επηρεάσει το προπολογισμό της Ένωσης και τα οικονομικά της. Ευχαριστώ. Η κυρία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή κύριε Επίτροπο, όσο και για το έγγραφο προβληματισμού. Πρέπει να πω ότι είχα κάπως υψηλότερες προσδοκίες σε σχέση με το περιεχόμενο του εγγράφου προϋπολογισμού. Ε, πρέπει να πω καταρχάς ότι μετά την ε, κοινοποίηση της Λευκής Βίβλου στα κράτη-μέλη ήταν παραπάνω από σαφές ότι η λύση δεν θα είναι κάποια από τα πέντε, αλλά ένα συνδυασμό ε, σεναρίων. Αυτό κατέστη σαφέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ε, τώρα συζητούμε για το μέλλον του νοσιακού προπολογισμού, αυτό θα πρέπει αμέσως να το λαμβάνουμε υπόψη. Εξού και περίμενα από τον Επίτροπο κάποιες προτάσεις για το πώς βλέπει τη διάρθρωση του προπολογισμού μετά το 2020. Πρώτα να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η νέα διάρθρωση και μετά να συζητήσουμε και όχι πάλι να συζητούμε βάση πέντε σεναρίων αφού ξέρουμε ότι ένα μείγμα τελικά σεναρίων θα ισχύσει σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού βάσει επιδόσεων. Αυτό είναι ένα στόχος Βέβαια θα πρέπει να διαβάσω ενδελεχώς ε, το έγγραφο συνολικά. Αλλά αν ε, διαβάσω το κομμάτι για τη συνοχή λέει ότι ότι ο στόχος είναι η ταχύτερη υλοποίηση και προβλέπονται μέτρα για την ε, πιο γρήγορη εκταμίευση που δεν έχει να κάνει όμως ε, με την ταχύτερη εφαρμογή. Το νη συν 1, συν 2, συν 3 είναι διαφορετικό. Πρέπει να είμαστε πιο ταχείς, άρα θέλουμε νέους κανόνες που θα αρχίσουν να ισχύουν ευθύ αμέσως από την έναρξη της επόμενης περίοδου για να έχουμε ταχύτερη εφαρμογή των πολιτικών συνοχής. Επίσης, ε, για αρκετό χρόνο ε, μιλήσατε για την προεντοξιακή ενίσχυση και επιγραμμίσατε, υπογραμμίσατε τη Σερβία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και άλλες χώρες και τη Βοστελεσικοβίνη να τις αναφέρουμε. Δεν ήταν φίλος πόλεμος. Είχαμε σερβική επίθεση κατά της Κροατίας. Κύριε Βαϊντέρ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριο Έτσιγκερ για τις προσπάθειές σας. Αντίθετα από τη συνάδελφο, θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό το έγγραφο, ήρθε την κατάλληλη στιγμή και πιστεύω βεβαίως ότι υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η κυρία Μάλετιτς μίλησε για την πολιτική της συνοχής, θα συμφωνήσω σε αυτό. Έχω και εγώ κάποιες ανησυχίες για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή. Εάν ε, από τα πέντε σενάρια καταλήξουμε σε ένα μόνο, το πέμπτο, με μια μικρή αύξηση στους σπόρους της συνοχής, τότε ισχύει μόνο το σενάριο 5 για μένα. Γιατί όλα τα άλλα προβλέπουν περικοπές για τη συνοχή και δεν θα ήταν σωστή επιλογή για την πολιτική μας αυτή. Επί παραδείγματι, και επειδή είμαι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο θα έλεγα ότι οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις ε, ολοκληρώνονται, πραγματοποιούνται καλύτερα μεταξύ κρατών που έχουν αντίστοιχο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό καθήκον που έχουμε αναλάβει, να βοηθήσουμε εκείνα τα κράτη τα οποία δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να ε, ενισχυθούν ακόμη, να αναπτυχθούν ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ταχύτερα για να φτάσουν στο επίπεδο αυτό. Η πρότασή σας για 5 συν 5 χρόνια είναι καλή, για μένα πολύ καλή, όπως και οι εισφορές των κρατών. Βεβαίως είναι επιφυλακτικοί οι συνάδελφοι, διότι δεν θα θελήσουν ίσως απαραίτητα να δώσουν πρόσθετη εισφορά τα κράτη, αλλά το επίπεδο ούτως ή άλλως δεν αντιστοιχεί στα, στις ανάγκες αυτά που έχουν υποσχεθεί δηλαδή τα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα να φτάσουμε σε μια αύξηση των ε, εισφερομένων στον προπολογισμό ποσό. Επίσης για το διοικητικό κόστο έχω ερώτηση, γιατί έχουμε 6% διαχειριστικό κόστο στι δραστηριότητε Δεν είναι αυτό υπερβολικό. Η μισθή, επί παραδείγματι, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, αυτά που πληρώνουν, έχουν πολύ ψηλού μισθού. Η κοινωνική ασφάλιση των υπαλλήλων επίση κοστίζει πολύ. Βλέπετε εκεί δυνατότητα για κάποια εξοικονόμηση πόρων. Ευχαριστώ. Ντονάνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όταν λέτε να περιοριστούν ε, οι επιστροφές θέμενη αξία, οικονομία κλίμακας. Βεβαίως πολύ καλά, αλλά πρώτα πρέπει να γνωρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε από κοινού τι πολιτική θέλουμε. Γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές, υπάρχουν και εθνικές, μπορεί να υπάρχουν και περιφερειακές πολιτικές. Επομένως θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αρμοδιότητες σε κάθε επίπεδο ε, πολιτικής δραστηριότητας. Να ξέρουμε τι κάνουμε από κοινού πριν διευκρινίσουμε τα δημοσιονομικά θέματα. Το ζήτημα των ιδίων πόρων ε, έχει ουσιώδη σημασία βεβαίω, και θέλω προσωπικώς να επίστησω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση αυτή να προχωρήσουμε στην προβολή κάποιων δημοσιονομικών μέσων τα οποία έχουν επιζήμια δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. διότι υλοποιούν πολιτικές όχι δημόσιες, αλλά ιδιωτικές, οι οποίες απλώς υποστηρίζονται από δημοσιονομικούς πόρους, από αυτά τα δημοσιονομικά μέσα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει τις δυνατότητες για επενδύσεις, αλλά να είναι και κατανοητό στο κοινό το τι κάνουμε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέλ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Είμαι συντονίστρια εκ μέρου τη ομάδα μου στην Επιτροπή Περιφερειακή Πολιτική. Θα σα ξαφνιάσω αν μιλήσω τη, για την πολιτική την περιφερειακή εδώ. Και πρέπει να πω ότι ακούγοντα τα διάφορα, βλέποντα μάλλον τα διάφορα σενάρια, αισθάνθηκα συντριβή, διότι ε, Χωρί να υπάρχει καν λόγο, εγκαταλείφθηκαν πολλέ από τι δυνατότητε και περίμενα ένα έγγραφο που μάλιστα συντάσσεται με την κυρία Κρέτσου από κοινού, το οποίο όμω θα έδειχνε πολύ πιο σαφή στράτευση υπέρ τη περιφερειακή πολιτική. Ήταν πολύ πιο εύκολο να ε, κοκκινήσετε ή να μαυρίσετε κάποια σημεία των ε, δραστηριοτήτων, αλλά ταυτόχρονα εγκαταλείπεται και μια αρχή που σημαίνει ότι κάθε ε, περιφέρεια μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την πολιτική συνοχή. Και αυτό συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή όπου η πολιτική της συνοχής είναι το μόνο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι κατανοητό για τον πολίτη, το οποίο έρχεται κοντά στον πολίτη και το οποίο του επιτρέπει να δει την άμεση διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και μόνο από μένα αποτελεί για, ε, για τα προγράμματα αυτά σαφή προσθεμένη αξία. Και σε αυτό πρέπει να υποστηριχθεί η πολιτική της συνοχής. Πιστεύω δε ότι πρέπει μαζί να καταφέρουμε να βρούμε δρόμους και τρόπους ώστε να μην εγκαταλείψουμε αυτές τις επιλογές και νομίζω ότι εάν μπορέσουμε να απλουστεύσουμε έστω ναι, αυτή την πολιτική ώστε να μην έχει το διαχειριστικό κόστος του 6% γιατί και αυτό μπορεί να είναι μια λύση είμαι διτεθειμένη να την επιδιώξω αλλά ταυτόχρονα να μην χαθεί η δυνατότητα της συμμετοχής για κάθε περιφέρεια, να μην χαθεί σε εποχές που εκφράζεται τόση επιφυλακτικότητα και δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να χαθεί η δυνατότητα για συμμετοχή όλων των περιφερειών στη συνοχή και δεί νομίζω ότι θα ήταν το χειρότερο από τα σενάρια αυτά. Ευχαριστώ. Νόβακοφ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχω μία ε, ευχή να πάρει το Όσκαρ ένα από τα πέντε σενάρια για να το καταφέρετε αυτό θα χρειαστείτε ε, την υποστήριξη των Ευρωβουλευτών. Και για να λάβετε το Όσκαρ για ένα από αυτά τα σενάρια θα πρέπει να τα αλλάξετε κάπως, να τα τροποποιήσετε. Συμφωνώ με την κυρία Κρέλ και προσθέτω θα, θέλετε, θα χρειάζεται και την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειακών θεμάτων, γιατί τα περισσότερα σενάρια προβλέπουν περικοπές στη συνοχή και στην, ε, πολιτική της γεωργίας. Και πώς θα το πούμε αυτό ε, στους λαούς μας όσο έχουμε το Brexit, όσο με σουρανή κρίση, μεταναστευτική, έχουμε την ε, οικονομική κρίση στην Ελλάδα και μπορεί και άλλες κρίσεις στο μέλλον. Φαντάζομαι όλοι θα σας υποστηρίξουν για να περάσουμε αυτή τη διαδικασία μαζί αλλά θέλω να μας διαβεβαιώσετε ότι θα είστε ανοιχτός, διαθέσιμος και συνεργάσιμος, διαλεκτικός στις διαπραγματεύσεις και όποιο σενάριο αν επιλέξουμε για προτεραιότητα, ως προτεραιότητα θα πρέπει να, να το τροποποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον και όφελος των συμπολιτών μας. Η κυρία Τομά, για μισό λεπτό. Καλώς. Μετά την φιλική πίεση που μου ασκήσατε, αποσύρω το έτοιμά μου για ε, να μιλήσω και πάλι. Ε, τότε θα υποφεληθώ εγώ ευχαριστώντας σας ε, για να θέσω και εγώ δύο σύντομες ερωτήσεις ε, στον Επιτρόπο. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή, την έκπτωση, μερικές χώρες θεωρούν ότι αν καταργήσουμε τι επιστροφές, μερικές χώρε θα εισφέρουν λιγότερο. Αν όμως καταργήσουμε τι επιστροφές, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες συνεισφορέ. Ε, δεν ξέρω, το περιμένουμε γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητες για τα έσοδα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ε, προοπτικές ε, αναθεώρησης των, του μηχανισμού των εσόδων και αν ε, έχουμε για παράδειγμα τα έσοδα από τις, εκπομ... τις δικαιωμάτων εκπομπών και προσθεθούν αυτά στον προπολογισμό θα είναι ένα πλέον έσοδο. Γίνεται επίσης, υπάρχει πιθανότητα μείωση ε, των ε, δαπανών τη ΚΑΠ. Η κοινή όμω γεωργική πολιτική έχει ω στόχο την εξασφάλιση γεωργικού εισοδήματο. Ε, την εξασφάλιση εισοδήματο στους γεωργούς. Οπότε, εγώ δεν είμαι υπέρ της, των περικοπών στην ΚΑΠ. Αν όμως χρειαστεί να κάνουμε κάποιες οικονομίες, μπορείτε να διανοηθείτε μία αναθεώρηση της εμπορικής ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση κάποιων ε, πολιτικών ελεύθερων συναλλαγών που χρησιμοποιούν ως ε, ανταλλακτικό μέσο μερικές φορές τη γεωργία. Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε την τιμή των γεωργικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να βελτιώσουμε το γεωργικό τους εισόδημα και να τους καταστήσουμε λιγότερο εξαρτημένους από τις ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, είναι δύσκολο να ε, προβλέψουμε δαπάνες σε κάποια κεφάλαια και πολιτικές αν ταυτόχρονα δεν ε, αναθεωρήσουμε κάποιους κανόνες που αφορούν τον ανταγωνισμό ή τις διαπραγματεύσεις για τις συνθήκες ε, ελεύθερου εμπορίου ή ελεύθερων συναλλαγών. Ε, συμφωνώ με τους ε, πέρους και τα με των συναδέλφων γιατί πραγματικά ήταν συναρπαστική ομιλία σας και τροφοδοτήσατε τη συζήτηση όχι μόνο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών αλλά και σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά και σας δίνω το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις για τις συστάσεις, για τις επικρίσεις. Να ξέρετε ότι οι γενικοί διευθυντές που είναι παρόντες καταγράφουν και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις. Πέντε ήταν οι επιλογές, τώρα έχουμε άλλες 25. Αρκετά ετερογενής η εικόνα, επαναλαμβάνω, αρκετά ετερογενής η εικόνα που μας δόθηκε. Πολύ σωστά όμως, γιατί είμαστε ακριβώς στις αρχές της συζήτησης. Σε 3,5 χρόνια και 3 μέρες ξεκινάει το μέλλον το δημοσιονομικό που συζητούμε. Δεν υπάρχει λόγος για ανυπομονησίες. Σε 3,5 χρόνια και 3 μέρες ξεκινάμε. Υποθέτω ότι το 5 συν 5 πρέπει να το κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και να προσδιορίσουμε και το δημοσιονομικό δίκαιο πιο προσεκτικά επίσης. Για τα 5 χρόνια. Τα αιτιολογείτε και πολύ σωστά με την πενταετή θητεία σας. Αλλά να σας πω εγώ, εγώ ως Επίτροπος που λύγει η θητεία μου τον Οκτώβριο του 19, πώς μπορώ να έχω απέτηση να προσδιορίσω τη δημοσιονομική πολιτική για την προσεχή δεκαετία. Και εσείς. Εάν βάλουμε λοιπόν ως συλλογισμό την παράλληλη διάρκεια μιας θητείας, με αυτήν του προϋπολογισμού, θα πρέπει κάθε κοινοβούλιο να έχει την ε, προοπτική να ορίσει μέχρι το 2026 το προϋπολογισμό. Όχι εγώ δηλαδή, όχι εσείς, ένα επόμενο κοινοβούλιο. Άρα αυτή η επιχειρηματολογία δεν στέκει πολύ. Ε, θέλω να πω, δεν στέκει απαραίτητα. Το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε περισσότερο. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σωστά. από τη διαδικασία της Λευκής Βίβλου ε, είμαι πεπισμένος, γιατί εκφράστηκαν σαφείς ε, ε, γνώμες υποστήριξη από τους προέδρους των πολιτικών σας ομάδων, είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι ήταν καλή επιλογή. Σεμινάρια ακούγονται, διατυπώνονται παρατηρήσεις κτλ. Ναι, βεβαίως τις λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά. Με το Brexit, ρωτάμε τι αλλάζει, πού πρέπει να προχωρήσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερες ταχύτητες προτεραιότητες, άλλα πράγματα πρέπει να εγκαταλειφθούν ενδεχομένως. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Και αυτά είναι και οι, προ... είναι και οι προβληματισμοί των πολιτών. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν βουλευτές που όντως είναι εκλεγμένοι και λένε θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Άλλοι πάλι λένε θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. κρατημέλη τα οποία υποστηρίζουν μια διακυβερνητικού τύπου διαδικασία νομοθετικής παραγωγής και μια Ευρώπη περισσότερων ταχυτήτων. Άλλα κρατημέλη τάσσονται κατά μια τέτοια επιλογή. Και η ιδέα μιας ε, πορείας η οποία θα είχε 20 μέλη στην πρώτη φάση για την εισαγγελία παραδείγματι και 8 εκτός. Πάλι δύο ταχύτητες είναι. Όλα αυτά τα λαμβάνω υπόψη και γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικό στα όσα διατυπώνω μέσα στο έγγραφό μου. Δεν προσπαθώ να καθοδηγήσω. Θα δείτε στους επόμενους μήνες θα γίνουν πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Ελπίζω να μην σας φανούν υπερβολικά συγκεκριμένες. Γιατί θέλω να υλοποιήσω τις ε, προσδοκίες. Όχι όλες όμως, γιατί ορισμένες εσκεμένα δεν θα τις ε, υλοποιήσω, δεν θα τις εκπληρώσω. Έχουμε χρόνο, έχουμε κάποιο χρόνο, θα τον αξιοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα του προβληματισμού, του αναλογισμού, της σκέψης, ε, της θεώρησης και της ακρόασης. πρέπει να αφουγκραστούμε ένας τον άλλον. Με την Πρατισλάβα ξεκίνησε μια διαδικασία που συνέχισε με τη Ρώμη δύο ευρωπαϊκά συμβούλια με ωραίες οικογενειακές φωτογραφίες ανεφετέρου. Ξέρουμε τι θέλουν και τι προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, Αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι αυτά είναι ένα σχέδιο ευρωπαϊκό και χρειάζεται περισσότερο χρήμα. 15 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Ε, έχω επισκεφθεί, έχω συναντήσει τους ε, υπουργούς τους. Πολλοί λένε καλύτερες δαπάνες. Ε, αυτό που λέμε στη Σουηδία είμαι οικονόμος, δεν δίνω παραπάνω χρήμα. Να κάνουμε οικονομία μόνο. Φεύγουν οι Βρετανοί, μας λείπουν 16%, 11 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα. Εμείς που μένουμε πίσω έχουμε πάντα το, το επίπεδο του 1%. Είναι ισχυρή αυτή η ομάδα. Και βεβαίω, αν θέλουν, μπορούν και στι χώρε του και στι ε, κυβερνήσει του, μέσω των κυβερνήσεών του μάλλον, να φέρουν κάποιε αλλαγέ. Ο κύριο Γκάιερ, λοιπόν, ο φίλο Γκάιερ, μου έστειλε μια επιστολή σήμερα που μου λέει ότι θα πρέπει να προσπαθήσω να πείσω και του ε, φίλου μου, του ε, πολιτικού, στο Βερολίνο και το Μόναχο. Θα κάνω, να δω, θα τα καταφέρω μόνο. Μα δεν χρειάζομαι όμω το Μόναχο, το Βερολίνο μόνο, την κυβέρνηση. Μα κύριε την ούτω ή άλλω στην αντιπολίτευση θα είσαστε, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, θα πείσω την κυβέρνηση, θα χρειαστεί μόνο την κυβέρνηση να πείσω από το Σεπτέμβριο και μετά. Αλλά, αλλά υπάρχει ανάγκη για στενέ επαφέ και θα αγωνιστώ για περισσότερα, για, για νέα μέσα. Σας ε, διαβεβαιώ με την ιδιαίτερη προσθεμένη αξία, με την καλύτερη αξιοποίηση, με το spending review, στην πολιτική συνοχής, βρίσκεται η πολιτική συνοχή σε μια κάποια κρίση. Εγώ προσπαθώ να εξασφαλίσω, ζητώ σταθερά κονδύλια για τη συνοχή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και οι περιφέρειες και τα κράτη θα αντλούν τους πόρους χωρίς καθυστερήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιδόσεις στην απορρόφηση από πλευράς των κρατών μελών δεν είναι πιστικές. Πού μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι περικοπές. Πολύ καλή ερώτηση. Εμείς ως Επιτροπή εφέτος είμαστε έτοιμοι με 5% λιγότερο προσωπικό και καλούμε και το Κοινοβούλιο την επόμενη χρονιά να παρουσιάσει την ίδια εικόνα. Περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένω. Τα τελευταία χρόνια πάγωσαν για δύο χρόνια οι μισθοί και κάναμε και πολλά άλλα και όντως και εγώ πιστεύω ότι κάθε υπάλληλο στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ίδια αμοιβή στο ίδιο κλιμάκιο και στον ίδιο βαθμό. Ο κάθε ένας. Ο κάθε ένας. Αλλά τότε δεν μπορώ να προσλάβω ούτε έναν Γερμανό παραπάνω. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας Γερμανός. Ε, μίλησα με τον Γκάμπριελ στο Βερολίνο, το Υπουργείο Εξωτερικών, για να πείσω υπαλλήλου να έρθουν σε έναν διαγωνισμό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι ε, από το κάθε κράτος μέλος να έρχεται ο καλύτερος, ο επιστήμονας, ο χημικός, ο οικονομολόγος, ο, αυτός που θα δει όμως μια θέση εργασίας ελκυστική για να πάει να τη ζητήσει. Όχι, σας, σας παρακαλώ, ελάτε μαζί μου, τόση γοητεία που έχετε, ελάτε μαζί μου στο Βερολίνο και πείστε τους... Ε, ε Γερμανούς, τους νεαρούς του Πότσδαμ, του Βερολίνου ε, ή του Μονάχου να έρθουνε. Εσείς ω γοητευτική Λουξεμβούργια θα τα καταφέρετε ίσως. Αλλά σα διαβεβαιώ ότι η βιομηχανία πληρώνει πιο πολλά. Η BASF, η Philips, η Bosch. Εμείς πρέπει να μπορούμε να διεκδικήσουμε όχι περισσότερους, τους καλύτερους. Τους καλύτερους να είμαστε ελκυστικοί ω εργοδότη. Βουλευτής, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Ελεγκτικό Συνέδριο, Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε ελκυστικό εργοδότη. Και αυτό το υποστηρίζω ανεπιφύλακτα. Ακούστηκε μια ερώτηση αν θα μένουν όλες οι περιφέρειες μέσα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως παραμένει αυτό στο έγγραφο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να χαθεί κάποια περιφέρεια. Αλλά το ζήτημα το θέτουν τα κράτη-μέλη και καποιοι ευφυει ευφύς οικονομολόγοι από ορισμένα κράτη-μέλη. Εγώ προ το αποτέλεσμα μαζί σα είμαι. Αλλά πρέπει να προωθηθούν οι πιο φτωχέ περιφέρειες και σε ένα έγγραφο προβληματισμού Πρέπει να διατυπώνουμε σαφείς θέσεις και όχι ανόητες που θα οδηγήσουν στην διαμόρφωση μιας σαφής πρότασης, μιας σαφούς πρότασης. Το lower share, χαμηλότερο ποσοστό, δεν σημαίνει τα less money, λιγότερο χρήμα. Το, εάν τα, ο, τα κονδύλια της συνομονοχής παραμένουν σταθερά, παραμένουν σταθερά ή παραμένουν της ε, και μετά θέλουμε να βάλουμε μέσα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και την αναπτυξιακή βοήθεια ή την άμυνα, τότε μπορεί το ε, ποσοστό, ο λόγος δηλαδή να μειωθεί, αλλά το ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες, του επόμενους μήνες. Η στρατηγική και το όραμα. Το όντι. Και παρατήρησε ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Κοιτάξτε, το έγγραφο προβληματισμού για την άμυνα που αναφέρεται σε 1,5 δις το χρόνο για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο για την άμυνα και την ασφάλεια. Εάν απορριφθεί, θα είναι πιο απλά τα πράγματα για τον προϋπολογισμό από ότι αν γίνει δεκτό. Γιατί φυσικά ένα τέτοιο ποσό επηρεάζει σημαντικά τον προϋπολογισμό προς τα πάνω ή προς τα κάτω εάν θέλουν οι Βρετανοί ας πούμε, να μείνουν ε, συνεργάτες, συνεταίροι στην αναπτυξιακή βοήθεια και κρατήσουν τη συμβολή τους στο Development Aid Fund, στο Ταμείο Βοήθειας για την Ανάπτυξη και συνεχίσουν να συνεισφέρουν, να συνεισφέρουν σε αυτό, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ποσό. Αν βγει πάλι πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και πάλι, αν μπει στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αυτό το ταμείο, έχει να κάνει με ενίσχυση και των προνομιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Βρετανοί για το 2019-2020 δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση. Ουσιώδη ζήτημα για εσά για το παρόν Κοινοβούλιο. Εάν αρνηθούν, εάν αρνούνταν οι Βρετανοί και οι διαπραγματεύσει για το διαζύγιο προχωρούσαν με το worst case σενάριο, τότε θα άλλαζε και η βάση δημοσιονομική και για το 2019 και το 2020, αλλά και για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο εκ βάθρων, γιατί θα μιλούσαμε για 100 δισεκατομμύρια 2019-2020, αλλά και παραπέρα θα λείπανε τόσα σημαντικά ποσά και γι' αυτό αυτή η σημαντική προκαταρκτική απόφαση πρέπει πρώτα να ληφθεί από τους Βρετανούς ή μαζί με τους Βρετανούς, για να συζητήσουμε την περίοδο για μετά το 2020. Στη γεωργική πολιτική, την κοινή γεωργική πολιτική, κοινοτικοποιημένη πολιτική της γεωργίας, βεβαίως και είναι πολύ σημαντική. Αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε χωρίς καμία περικοπή σε αποτελέσματα, διότι δεν πρόκειται κανείς να μας υποστηρίξει. Και θα ήθελα να πω επίσης, σε σχέση με τις ε, συγκρίσεις. Εσείς έχετε και πιο πολύ εμπειρία βέβαια από ό,τι εγώ. Στην πρώτη τελευταία ε, δημοσιονομική περίοδο είχε κάνει πολύ συγκεκριμένε προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έριξε μια ματιά το Συμβούλιο, πλουφ, στο κάλαθο των αχρήστων και δεν υπήρχε πλέον πρόταση. Ο Μπαρόσο και Λεβαντόφσκι είχαν μία πρόταση μετρημένη, ρεαλιστική, απερίφθη όμως. Και από την πρώτη μέχρι τελευταία μέρη, η μέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ό,τι μπορούσε για να προχωρήσουν αυτά τα... Τα... αυτές τις προτάσεις. Ας το δούμε λοιπόν με τα μάτια ανοιχτά. Πολλά κράτη-μέλη δεν μας λένε τι δίνουν, τι μπορούμε να περιμένουμε. Κάποιοι έχουν μπροστά τους προεκλογική περίοδο από ένα χώρο γερμανόφαινο θα έλεγα παραδείγματι, ότι ακούγεται ότι θέλουν να περικοπούν στο ίμιση οι, ε, και ότι δεν πρόκειται να δώσουν πια κανένα τάλαρο στον προϋπολογισμό πέραν αυτού. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. στη γεωργική πολιτική. Θα ξεχωρίσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Θα τις αναφέρουμε κάπου ρητά. Εγώ είμαι ε, σε αυτό το θέμα. Προέρχομαι από χώρα με μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Άρα μπορούμε να το συζητήσουμε με βάση και τις πραγματικές ανάγκες, αλλά να κοιτάξουμε ίσως και μια σταδιακή μείωση ανά εκτάριο, παραδείγματι. Είναι κάτι το οποίο μέσα στη διαδικασία αυτή του προβληματισμού πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό και αποδεκτό αποτέλεσμα. Πολλά είναι τα εκκρεμή ερωτήματα. Σήμερα ξεκινούμε, σήμερα δίνουμε το εναρκτήριο λάκτισμα. Ε, περιμένω τις προτάσεις σας. Είμαστε εδώ τις επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτές τις ακατέργαστες προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα διαμορφώσουν τελικά το τελικό αποτέλεσμα. Ίσως με την τρέχουσα επιτροπή, πάνω απ' όλα μαζί με εσά, μαζί με το ε, τωρινό κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Οπότε θα περάσουμε ένα πολύ μελετηρό καλοκαίρι θα αναλύσουμε διεξοδικά το έγγραφο που μας υποβάλλατε. Μας είπατε θα προσπαθήσετε να πείσετε και τις κυβερνήσεις. Και αν κατάλαβα καλά, είναι πιο εύκολο να πείσετε τις κυβερνήσεις ε, μετά <laughs> το Σεπτέμβριο. Είπατε ότι μετά το Σεπτέμβριο θα είναι πιο εύκολο να πείσετε τις κυβερνήσεις. Οπότε αν θέλουμε να πιστούν οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να τις ενθαρρύνει γι' αυτό η κοινή γνώμη. Οπότε θα πρέπει εμείς να τροφοδοτήσουμε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι δημόσια αγαθά μπορούν να έχουν διαχείριση σε εθνικό επίπεδο και άλλα λόγω παγκοσμιοποίησης μπορούν να μόνο να κανονιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν το αποφασίσουμε αυτό θα πρέπει να αντιλήσουμε και κάποιες, κάποια συμπεράσματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο, τους συζητητές. Οι συντονιστές θα συνεδριάσουν αύριο στις 8.30 και η Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 10. Λύεται η συνεδρίαση.